Σίγουρα αυτή η εφαρμογή ε, θα διέπεται στο μέλλον από τους, ε, σίγουρα από τους ελέγχους τους οποίους προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα της Ουγγαρίας αλλά ταυτόχρονα και θα διέπεται αυτή η εφαρμογή και από την δράση των υπερεθνικών οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν ε, μπορώ να γνωρίσω όμως αυτό που άκουσα σε ό,τι αφορά την προστασία των μειονοτήτων στο, στην, ε, στο Σύνταγμα της Ισπανίας ε, όπως επίσης και τα σχόλια για άλλα συντάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Σύνταγμα της Ισπανίας δεν υπάρχει κανενός είδους σκιά διάκρισης ε, με βάση το φύλλο, με βάση την εθνοτική καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλη. άλλο κριτήριο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Ουγγρικό Σύνταγμα, αλλά ε, η αλήθεια είναι πως ε, σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο πολλές φορές ακούστηκε η άποψη ότι το Ουγγρικό Σύνταγμα θα πρέπει να εξασφαλίζει την πολιτική πολυφωνία και την δυνατότητα εναλλαγής πολιτικών στην διοίκηση του κράτους. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των φιλελευθέρων, ε, κυρία Βέιμπερ, για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το νέο θεμελιώδες νομοθετικό κείμενο της Ουγγαρίας, που θα έλεγε κανείς ένα αμφιλεγόμενο κείμενο για να είναι σύνταγμα, έχει τρέξει μέσα σε ένα μήνα όλες τις διαβουλεύσεις και η Επιτροπή της Βενετίας